Good morning, ladies and gentlemen. Welcome in Καλημέρα σας. Ε, σας καλωσορίζω σε αυτή την αίθουσα που δεν συνηθίζουμε να συνεδριάζουμε. Δεν σας βλέπω καν εδώ, τέλος πάντων. Γεια σας. Θα προσπαθήσω να σας αναγνωρίζω. Τέλος πάντων, ε, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να αρχίσουμε την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ΡΕΤΖΙ. Έχετε μπροστά σας την μερίσια διάταξη. Συμφωνείτε να εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης, κύριε Βανίστερο. Ευχαριστώ. Ε, μπορώ ε, να δεχτώ την, ε, το σχέδιο μερίσης διαταξής. Αλλά δύο ερωτήσει έχω. Η κυρία Κρέσου για λυμμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να έρθει. Ζητάει να το συζητήσουμε το θέμα την επόμενη φορά, μα γίνεται. Και μετά. Έχουμε το, να δούμε το νέο Γενικό Διευθυντή, για να το γνωρίσουμε καλύτερα. Έχουμε και τη σύσκεψη των συντονιστών σήμερα. Λοιπόν, για τις ε, επόμενες ε, ημερησίες διατάξεις καλό θα ήταν να σκεφτούμε το ενδεχόμενο ε, σύνταξη ψηφίσματος προς την Ολομέλεια από την Επιτροπή Ρέτζη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, συμμορφωθούν με την εξάντερη σημότητα μέχρι το τέλος του χρόνου. Και όσοι δεν ε, καταρτήσουν εθνικές στρατηγικές μπορεί και να χάσουν τη χρηματοδότηση για την τρέχουσα περίοδο. Έχει κέρια σημασία το ζήτημα λοιπόν. Για να προετοιμάσουμε και την ψηφοφορία για αυτό το ψήφισμα πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία και στις αρχές του 17 στην Ολομέλεια πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποια θέση θα τηρήσουμε. Οπότε, ε, μήπως ε, οι πολιτικές ομάδες να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα αναλάβει την πρωτοβουλία και εκείνη θα ε, χαράξει πορεία και θα αναπρογραμματίσει τη χρήση των κονδυλίων. Πρέπει να δούμε για αυτή την ε, περίοδο αυτά τα 360 δισεκατομμύρια το κονδύλι που έχουμε να δαπανίσουμε, αν δεν υπάρξει απορρόφηση τα πρώτα τρία χρόνια, θα πρέπει διακομματικά ίσως να προετοιμάσουμε καλά εδώ στη Ρέτζη την, ε, το δρόμο που θα προτείνουμε. Δεν το λέω για σήμερα, αλλά για να προγραμματίσουμε για επόμενες συνεδριάσεις ανταλλαγή απόψεων. Το ΕΛΚ έχει προετοιμάσει ήδη ένα σχέδιο, τέλος πάντων να ε, συνεργαστούμε όλοι. Και περίμενα να έρθουν όλοι οι δικοί μου, γι' αυτό μίλησα τόση ώρα. Ευχαριστώ, ίσως αυτό οφείλεται στην αίθουσα. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε σχεδόν ε, σχετιζόταν με τη μερίσια διάταξη αυτό που είπατε. Εγκρίνεται το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Θα δούμε τι θα γίνει με τις μελλοντικές συνεδριάσεις. Ανακοινώσεις της Προέδρου, δεύτερο σημείο. Ε, για να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα έχω ανακοινώσει ε, αποστολή στην Ελλάδα από τις 18 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Πριν από τρεις εβδομάδες επισκεφθήκαμε την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 11 συνεδριάσεις ε, κάναμε σε διάφορα επίπεδα πολιτικών αρχών. Ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Δραγασάκη, με τον κύριο Αλέξη Τσερίδα, Υπουργό Οικονομίας και διάφορους άλλους ηθήνοντες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Α, και με το Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκη και τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Αθηνών. Ε, επίσης έχουμε, ε, συναντηθήκαμε με τον συναδέλφους από την αρχή υποστήριξη των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων Συζητήσαμε για διάφορα ενδιαφέροντα προγράμματα, και κάποια αμφιλεγόμενα, το μετρό στη Θεσσαλονίκη και κάποια επιτυχημένα στον Πειραιά, αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε, η γραμματεία προετοίμασε ήδη την έκθεση και σας την έχει μοιράσει. Και είναι Υπάρχουν αντίτυπα μέσα στην αίθουσα αν ε, δεν το έχετε πάρει. Ήταν επιτυχημένη η αποστολή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η έκφραση αποστολής. Δυστυχώς ε, δεν φαίνονται καλά οι φωτογραφίες όταν τις τυπώνουμε. Δύσκολα να γνωρίζει κανείς τα πρόσωπα. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να βάζουμε περισσότερες φωτογραφίες στις εκθέσεις πολύ θετική επίσκεψη. Αυτό ήταν το βασικότερο. Περιμέναν περισσότερα προβλήματα, δυσκολίες και οι εκπρόσωποι των διαφόρων ε, πολιτικών αρχών σε διάφορα επίπεδα εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν να εργάζονται και να ε, δώσουμε το παράδειγμα με τη δουλειά που κάνω για τα διαρθωτικά ταμεία. Όταν έχουμε χρόνο ή όταν θέλετε μπορούμε να ξανασυζητήσουμε αυτή την αποστολή. Δεύτερη ανακοίνωση. Ετήσια έκθεση ε, συνεδρίαση Κοτέρα αύριο το απόγευμα θα λάβει χώρα συνεδρίαση από τις 2.30 μέχρι τις 5. Στη, φυσικά στο κτίριο της Επιτροπής των Περιφερειών. Είναι μία από τις εκδηλώσεις ε, σε αυτή την τρέχουσα εβδομάδα των περιφερειών εδώ στις Βρυξέλλες. Η εναρκτήρια συνεδρίαση ήταν ε, χθες, έγινε χθες στο, στο ε, ημικύκλιο, στο κοινοβούλιο. Ο κ. Βανιστερό ήταν εκεί. Νομίζω από πλευρά τη Επιτροπή των Περιφερειών θα είναι ιδιαίτερα συγκινητική η ευριανή συνεδρίαση και έχουμε και διάφορε προσδοκίε. Θέλει η Επιτροπή των Περιφερειών να λάβει γνώση των ε, προθέσεων του Κοινοβουλίου για την ε, περίοδο μετά το 2020, για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τρίτη ανακοίνωση 28 Σεπτεμβρίου είχαμε μια εκδήλωση οργανώσει στην αντιπροσωπεία της Βαβαρίας με τίτλο «Ανανεωμένη ισχυρή περιφερειακή πολιτική για όλες τις περιοχές μετά το 2020». Και πριν τη δεξίωση έγινε διάσκεψη για τη διαχείριση του μέλλοντος από τις περιφέρειες και όπως σας είπα διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών. 332 ερετοί από περιοχές από 32 κράτη-μέλη και 5 διαπεριφερειακές οργανώσεις υπέγραψαν κοινή δήλωση ζητώντας ε, κατοχήρωση της διατροτικής πολιτικής ε, μετά το 2020 από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ο κύριος Μάρκουλε, η κυρία Κρετσού, ο πρέσβης Πέτρη Γιάβουτσικ από τη Σλοβακική Προεδρία έλαβαν το βιβλίο υπογραφών και εγώ με την ιδιότητα μου της Προέδρου Α, σας δείχνω εδώ το TTP, τι έλαβα. Είναι αυτό το βιβλίο υπογραφών, πολύ βαρύ, πολύ εντυπωσιακό. Σας είπα 332 ερετή υπέγραψαν θα το δώσω στη γραμματεία ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο και σε εσά. Μπορείτε να δείτε ε, από τις χώρες σας ποιες περιοχές υπέγραψαν αυτή την κοινή δήλωση που είναι αρκετά ισχυρή στόχοδετημένη και σχετίζεται με το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Παραδίδει το βιβλίο στη γραμματεία λοιπόν. Έχω κι άλλη μια ανακοίνωση. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο το Σώμα των Επιτρόπων και η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συνεδρίασαν για να συζητήσουν ε, το πρόγραμμα εργασιών ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017. Σε κλάστες ε, οργανωθήκαμε όπως πέρσι, σε ομάδες δηλαδή. Είναι καλύτερος τρόπος αυτός για να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουν σε δύο ομάδες, μία για το πολιετές δημοσιονομικό και μία για τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Στην πρώτη, συμπροέδρευε πρώτη η Πρόεδρος Επιτροπής και και Επίτροπος Έτιγκερ, διότι η Αντιπρόεδρος Γεωργίευα δεν ήταν παρούσα τότε, εκείνη τη στιγμή. Στη, στη δεύτερη συμπρόεδρος ήταν ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και ε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ήμουν ε, για την δεύτερη ομάδα υπεύθυνη για τις δηλώσεις και συζητήσαμε την πολιτική συνοχή, τα διορθωτικά ταμεία και την επενδυτική πολιτική και τονίσαμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των διαστατικών ταμείων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την ανάπτυξη στην Ευρώπη ε, ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Πολιτικής. Ιδού, ολοκληρώνω έτσι τις ανακοινώσεις μου. Και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. σήμερα θα ψηφίσουμε για μία έκθεση και μία γνωμοδότηση που τροποποιεί το, ε, τροποποιεί το κανονισμό 1303 το 2003 για κάποιες διατάξεις σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση για κάποια κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με την χρηματοοικονομική του σταθερότητα, τεράστιος αυτός ο τίτλος. Αυτή η νομοθετική πρόσφαση σχετίζεται με το άρθρο 24 και για ε, άρθρο 120 παράγραφος 3 των, του κανονισμού δινών διατάξεων βάσει των οποίων επιτρέπεται συγχρηματοδότηση για τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ε, προτείνει η Επιτροπή να παραταθεί η περίοδος ε, όπου είναι πιθανή αυτή η χρηματοδότηση. Η τροπολογία για το άρθρο 24 αφορά κυρίως την Ελλάδα και για το άρθρο 120, ε, εδάφιο 3, την Κύπρο. Μου ζητήθηκε να είμαι εισηγητής για την Επιτροπή. Επί της αρχής την περασμένη φορά αποφασίσαμε χωρίς τροπολογίες να εγκρίνουμε την, απόφαση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Κορεπέρης στις 21 Σεπτεμβρίου αποφάσισε να εγκρίνει επίσης χωρίς τροπολογίες την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δύο συμβουλευτικές επιτροπές, η ΕΣΥ, η Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή και οι ΟΚΕ έχουν εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, ε, η... καμία από τις επιτροπές που συνέταξαν γνωμοδότηση δεν υπέβαλαν τροπολογίες. Ο πρόεδρος υποστηρίζει την προσέγγισή μας με επιστολή που απέστειλε. Είναι πάνω από 10 οι επιτροπές ε, που ε, γνωμοδότηση, που αποφάσισαν να μην συντάξουν γνωμοδότηση. Ε, μία ε, ενιαία ψηφοφορία λοιπόν για αυτή την ε, υπόθεση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Όχι. Ε, βγήκε αποτέλεσμα. Μπορέσατε να ψηφίσετε. καλό. Δεν δουλεύει το μηχάνημα. Συγγνώμη. Θα κλείσουμε την ψηφοφορία. Δεν ξέρω. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Ε, δουλεύει τώρα. Α, έχετε πρόβλημα. Να έρθουν οι τεχνικοί παρακαλώ. Δεν δουλεύει. Ε, μάλλον θα επαναληφθεί η ψηφοφορία. Ναι. Ψηφίστε τώρα παρακαλώ και πάλι. Όλα ψήφισαν όλοι. Ωραία. Κλείνει η ψηφοφορία. Ωραία, εγκρίθηκε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. 34 ψήφισαν ή 31 υποστήριξαν. Ε, να απόφαση 31 μέλη ψήφισαν υπέρ. Περνάμε τώρα στην ε, Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για το Κοινοβούλιο. Η συγκήτριά μας είναι η κυρία Μπρέσο. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Καλά. 96 τροπολογίες είχαμε. Έχουμε διάφορες ε, συμβαστικές. Είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Ε, συμβαστική 1 ε, υπέρ. Κατά. Αν και αποχές, ξέχασα. Όχι, ωραία, εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε έναν έλεγχο ηλεκτρονικό. Παρακαλώ, δυσκολεύομαι σε αυτήν την αίθουσα να καταλάβω πώς έχει κατάσταση, γιατί 14 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ήθελα επαλήθευση γιατί δεν μπορώ να... δεν τα καταφέρνω σε αυτήν την αίθουσα. Κύριε ε. μπορείτε να μετρήσετε εσείς τα μέλη του ΕΛΚ. Γιατί έχουμε έναν υπεράριθμο από εσά είναι. Ε, ένα από τα μέλη λοιπόν θα βγει, οι υπόλοιποι θα παραμείνουν, λέει ο κύριος Νίστελόι. Καλώς, η 15 θα πάμε στο δεύτερο τμήμα της. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Καλώς, να ελέγξουμε. Για το δεύτερο τμήμα της 15. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 16. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται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 The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίες. Απορρίπτεται, νομίζω, λέει η πρόεδρος. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46. Υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε καλώς για την 46 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρασε και απορρίπτεται Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω λέει ο πρόεδρος θέλετε να ελέγξουμε την 62 παρακαλώ άρχεται η ψηφορία της 62 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η ε, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 87 παρακαλώ Πέρας. Απορρίπτεται. «88 έως και 91 ταυτόσημες. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνονται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι, εγκρίνονται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Στο συγγνώμη λέει Α, Αχα, καταπίπτει. Μάλιστα. Σημαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται και Τώρα πάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του συνόλου. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32 ψηφίσαντες, 28 υπέρ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τώρα την ψηφοφορία, τις ψηφοφορίες. Και πάμε στο επόμενο σημείο. που είναι η ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική με συντάκτη τον κύριο Νίλσον ε, είπατε εκπρόσωπος ε, δημοσίευσε μια έκθεση με ακριβώς αυτόν τον τίτλο τον Απρίλιο οι επιτροπές ΑΦΕΤ και ΕΝΒΙ προχώρησαν σε γνωμοδότηση πρωτοβουλίες με βάση τον κανόνα 55. Παρακαλώ όμως ησυχία, αν έχετε σημαντικές συζητήσεις, παρακαλώ εκτός της αίθουσας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλσον λοιπόν έλεγα θα παρουσιάσει το σχέδιο εκθέσεώς του για τα βασικά περιφερειακά συστατικά της ε, προσέγγισης της στρατηγικής της Αρκτικής. Μέχρι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 5.30 είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε 2 Νοεμβρίου. Ο κύριος Νίλσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί που μου αναθέσατε το ρόλο του εισηγητή για τα θέματα Αρκτικής. Ε, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι καθήλυν αρμόδια, το ίδιο και, ε, και στην αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως και εμείς. Ε, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, έχει, φυσικά θα πρέπει να συντάξει γνωμοδότηση γιατί αλλιώς θα είναι λυπής ε, η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται εδώ μόνο για ασφάλεια, για εξωτερικές υποθέσεις, για το περιβάλλον, διότι σε αυτές τις περιοχές δεν βλέπουμε μόνο γάδο και πολικές αρκούδες, μένουν και άνθρωποι εκεί πέρα. Ε, και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό περιλαμβάνεται και η Γρυλανδία και η Βόρεια Ευρώπη. Έχουν μια καθημερινή ζωή ακριβώς όπως και εμείς. Προσπαθούν να δημιουργούν βιώσιμες κοινωνίες, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και γι' αυτό είναι το σημαντικό να δώσουμε και εμείς τη δική μας διάσταση, την περιφερειακή διάσταση στην όλη διαδικασία η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και με χώρες πέρα από τα εξωτερικά μας σύνορα και χώρες της Αρκτικής έχει ιδιαίτερη σημασία και φυσικά θα πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση που προβλέπεται ήδη για την εδαφική συνεργασία. Ε, θέλουμε επίσης να γίνει μέλος του Αρκτικού Συμβουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση με παρατηρητή είναι πάρα πολύ μεγάλο το ειδικό βάρος των διαρθρωτικών ταμείων για την ε, δημιουργία ανάπτυξη και θέσεων εργασίας στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν και μόνιμα ε, μειονεκτήματα φυσικά που έχουμε διαπιστώσει στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφέρειες, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ε, τι ε, χρειάζονται, όχι μόνο για τις δικές τους περιοχές, αλλά και για θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Δεν είναι πολυπληθείς οι περιοχές, όμως έχουν πολύτιμες γνώσεις που θα, ε, που θα έπρεπε να μοιραστούμε και εμείς για αυτά τα ζητήματα. Στι μελλοντικέ μα εργασίε, λοιπόν, θα πρέπει να ακούσουμε τι απόψει αυτών των περιοχών. Επίση, ε, η έρευνα που γίνεται στην περιοχή θα πρέπει να ενισχυθεί. Δεν πρόκειται μόνο για την οικονομία, αλλά και για τον ε, αγροτουρισμό, για το περιβάλλον, ε, για τεχνογνωσία. Ε, είναι πολυάριθμες οι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα εξεκέλευση τεχνολογίες σε αυτή την περιοχή και ε, νομίζω θα πρέπει να το τονίσουμε από πλευρά της Επιτροπής μας. Υπάρχει και μια παλιά πρόταση να συσταθεί ένα κέντρο για πληροφορίες για την αρκτική περιοχή στο Ροβανιέμι στην Φινλανδία. καλό θα ήταν να ακολουθήσει, να εγκρίνει αυτή την πρόταση και να συγκροτήσει αυτό το κέντρο ε, στο με μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπρεπε να την ενθαρρύνουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η περιφερειακή διάσταση που νομίζω θα έπρεπε να προσθέσουμε στην ανάλυση που θα κάνουν οι δύο συναρμόδιε επιτροπές. Αν έχετε κι εσεί άλλε προτάσει ε, με τα χαρά να τη λάβω υπόψη και να καταλήξω στο τελικό σχέδιο που θα υποβάλω στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νίλσον. Θα δώσω το λόγο στους Κιώδης, πρώτα απ' όλα. Ο κύριος Σκέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι διαμεσολαβητής μεταξύ της Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων και Περιφερειακών Υποθέσεων, όπου είμαι αναπληρωτής αλλά με χαρά να υποστηρίξω τον συνάδελφο Νίλσον γιατί νομίζω ότι είναι από τα βασικότερα σημεία εδώ είναι να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντικό είναι για την ε, αρκτική περιοχή η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία η οποία θα πρέπει να συνεχίσει όταν θα ολοκληρώσουμε το πολιετές ε, δημοσιονομικό πρόγραμμα ως το τέλος της δεκαετίας. Το ΕΛΚ επίση θα μπορούσε να υποστηρίξει την ιδέα, το σκεπτικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετάσχει ως πλήρης παρατηρητής στο Συμβούλιο για την αρχιτεκτονική. Αυτό που χρειάζεται και το λέγει το σχέδιο κειμένου είναι συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων, των τοπικών κυβερνήσεων, διότι είναι σημαντικό να έχουμε συνεχές ε, feedback από τους φορείς αυτούς που εργάζονται εκεί επί τόπου. Επίσης, η καινοτομία είναι πολύ σημαντική για την περιοχή της Αρκτικής η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει το έλλειμμα ανθρωπίνων πόρων και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και τόμα πρότυπα επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Εκ μέρους της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα έλεγα ότι ε, δεν μπορεί να βλέπουμε την Αρκτική μόνο ως περιοχή φίλων κρατών μελών και εταίρων. Πρόκειται για γεωπολιτική περιοχή με στρατηγικά συμφέροντα που συγκρούονται μεταξύ τους ενεργειακά, μεταφορικά και άλλα. Η, περιφερειακή πολιτική λοιπόν στις ε, συνοριακές περιοχές δεν είναι απλώς θέμα περιφερειακής πολιτικής. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μια εξωτερική διάσταση. Και ε, θα ήθελα να υποβάλω κάποιες παρατηρήσεις προς την κατένση αυτήν. Όπως τα γνωρίζετε, η Ρωσία είναι πολύ σημαντικός παίκτη στο πεδίο της αρτικής και πρέπει ρεαλιστικά να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο καταπατά την διεθνή νομοθεσία. Και τέλος, θα μου άρεσε η δημιουργία ενός κέντρου πληροφορίας στη Φιλονδία, προερχόμενος από την Εστονία, ε, που δεν είναι τόσο κοντά στην πιστεύω ότι οι Εστονοί θα μπορούσαν να υποστηρίξουν απολύτως τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στην γείτονα Φιλανδία. Ο κύριος Λιούαρ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και καλημέρα στους συναδέλφους αυτό το... στην ασυνήθιστη αυτή αίθουσα. Ε, να τονίσω ότι η ομάδα ECR με, τους, ε, με τα φιλανδικά και δανικά μέλη της είναι υπέρ του φόρουμ και της δικτύωσης και συνεργασίας για την ανάπτυξη δυνατοτήτων την επίγνωση των ε, δημοσιονομικών πόρων και των διεθνών αναπτυξιακών έργων. Εμείς ε, συστήνουμε στην Κομισιόν να προγραμματίσει εντός των υφισταμένων πόρων την ολοκλήρωση μέχρι το 17 της πρώτης φάσης που έχει προβλέψει μαζί με τις διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς που υπάρχουν και που εκπροσωπούνται σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις που είναι παρούσες στην Αρκτική και μαζί με τη Δανία, Σουηδία και Φιλανδία ως πλήρη μέλη, το ECR θα συνιστούσε σεβασμό για τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών αυτών μελών μαζί με τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Συμβουλίου της Ακτικής ως βασικούς φορείς εντός του, της περιοχής. Αναγνωρίζουμε ότι παρέχουμε χρηματοδότηση προς τις απόμακρες περιοχές, αλλά οποιοδήποτε υποστηρικτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ήταν αντικατάσταση των κρατών μελών, αλλά ακριβώς συμπληρωματικός. Επίσης αναγνωρίζουμε την κρίσιμη σημασία του Συμβουλίου της Ακτικής και της όλης περιοχής ως μοναδική περιοχή επιστημονικής σημασίας και ιδιαίτερα σχετικά με την έρευνα που διεξάγεται για την κλιματική αλλαγή. Η χρηματοδότηση αυτής της έρευνας θα είναι πολύ σημαντική. Θεωρούμε επίσης ότι οι φυστάμενες δομές και σχέσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται πλήρως. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε 200 εκατομμύρια ευρώ για υφιστάμενα ακτικά έργα μεταξύ του 6ου και 7ου ε, πλαισίου και εντός του ορίζοντα 2020 που όπως γνωρίζει η συνάδελφοι έχει διάφορους μη Ευρωπαίους συμμετέχοντες ε, θα πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να συνεργαστεί με όλους αυτούς τους φορείς και να συλλέξει κάποια, κάποιες εμπειρίες και συμπεράσματα. Ε, επίσης ε, υποστηρίζουμε να ολοκληρωθεί το κέντρο στο Ρόβανιέμι εντός χρόνου και εντός της δυνατότητας των πόρων που έχουμε. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, ίσως μπορώ να χρησιμοποιήσω και τη μητρική μου γλώσσα τα φινλανδικά διότι με την καλύτερη προετοιμασία αρθρώνεται η φωνή της Φινλανδίας σε σχέση με αυτά. Συνεχίζω φινλανδικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. <clears throat> Θα ήθελα εξ ονόματος της κοινοβουλευτής ομάδας ALDE να ευχαριστήσω πρώτα τον συνάδελφο Γιένς Νίλσεν για το καλό κείμενο το οποίο εξεπώνησε. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ισόρροπου πλαισίου όπου θα μπορέσει να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι θετικό ότι η πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με την Αρκτική αναγνωρίζεται εδώ έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία για τις ακτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσές, μικρομεσές επιχειρήσεις. Το δικό μας ταμείο αρρωγής υποστηρίζει με ιδιαίτερο τρόπο τον χώρο, την περιφέρεια της Ακτικής και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Η σπουδαιότητα αυτών των ταμείων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διαθέτουν κονδύλια με πολύ σημαντικό τρόπο η πληροφόρηση και η ανταλλαγή πληροφοριών θα ήταν καλύτερη. Θα έπρεπε εδώ σε σχέση με την Αρκτική να μην αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ξεχωριστά και να μην βλέπουμε μόνο τα προβλήματα του δικού μας τομέα. Η δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας λοιπόν είναι μια πολύ καλή δυνατότητα για μας να μπορέσουμε να ασκήσουμε την επιρροή μας και να βελτιωθεί η κατάσταση της Αρκτικής. Το οικοσύστημα της Αρκτικής είναι μοναδικό και προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες ε, και δυνατότητες και αν με καλό τρόπο σχεδιάσουμε τα πράγματα αρκετά προτερήματα θα μπορέσουμε να πετύχουμε αν η έδρα μόνιμα θα μπορούσε να βρίσκεται στο Ροβανιέμι τότε θα μπορούσαμε με πολύ καλό τρόπο να δράσουμε και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την Αρκτική να συλλέγονται εκεί. Η σημερινή κατάσταση είναι δυσχερής αλλά η βόρεια διάσταση της Αρκτικής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Θα είναι ένα φόρουμ συζητήσεων συζητήσεων λοιπόν με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ακόμα και σε σχέση και με τη Ρωσία. Θα μπορούσαμε να δώσουμε συνέχεια σε θέματα που είναι πολύ σημαντικά όπως τα θέματα της απόδοσης, αποδοτικότητας ενέργειας και των εταιρικών σχέσεων και η συνεργασία στις μεταφορές επίσης είναι πολύ σημαντική υπόθεση αυτή τη στιγμή το πώς λειτουργεί η βόρεια διάσταση περιορίζεται από τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Όμως παρόλα αυτά σε ένα συγκεκριμένο έστω μικρότερο πλαίσιο αυτή η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί. Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι ο Νίλσον ο συνάδελφος εξεπώνησε ένα εξαιρετικό κείμενο έκανε μια πολύ καλή έκθεση θα γίνει μια εξαιρετική έκθεση και ευελπιστώ ότι με βάση ακριβώς αυτή την έκθεση θα μπορέσουμε σχετικά σύντομα να μπορέσουμε στην πιο όμορφη πόλη της Ευρώπης Ροβανιέμι να έχουμε αυτή την έδρα. Σας ευχαριστώ. Ο Σκιώδης εισηγητής στη συνέχεια κύριος Κοσλέκα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης για μια πολύ καλή δουλειά που επετέλεσε. Συμφωνούμε με τις περισσότερες προτάσεις και στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό για την απασχόληση στην Αρκτική. Πρέπει να σκεφτούμε και τα θέματα της αηφορίας. Η αηφορία στην ανάπτυξη και η αηφόρος απασχόληση πρέπει να είναι τα θεμέλια για την ανάπτυξη του χώρου της Αρκτικής. Αυτοί, αυτές οι αρχές θα πρέπει να αναπτυχθούν και να μετεξελιχθούν όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία και ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να επικεντρώνονται υπό το πρίσμα αυτό όπως ε, αρθρώνεται σε αυτή τη γνωμοδότηση η δημιουργία φιλόδοξων στόχων για την αηφορία στην ανάπτυξη δεν είναι εφικτή αν δεν δώσουμε την δέουσα προσοχή στην ποιότητα της διαχείρισης διότι πρέπει να εμπλέκονται οι τοπικές κοινότητες στις λήψεις αποφάσεων και στην εκτέλεση. Η συνεργασία λοιπόν των τοπικών αρχών, δήμων, κοινοτήτων και λοιπόν είναι αναγκαία δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε διότι οι τοπικές αρχές στο περιφερειακό επίπεδο γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα και ξέρουν τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Αν δεν εμπλακεί σε αυτό το επίπεδο λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα τα καταφέρουμε. Να στρέψουμε μεγαλύτερη προσοχή στη συνεργασία των περιφερειών στον χώρο της Αρκτικής. Να ξεκινήσουμε με τη διαμεθοριακή συνεργασία. Να δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του ιδιαίτερα ευάλωτου κλιματικού παράγοντα που υφίσταται τα πλήγματα των κλιματικών κλιματικών αλλαγών έτσι θα πρέπει να συνεισφέρουμε για την αηφόρο ανάπτυξη και στην ευρωπαϊκή πλευρά της Ακτικής αλλά και στην απέναντι πλευρά της Ακτικής. Πρέπει να συνεισφέρουμε έτσι συνολικά στην πολιτική για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μπορεί με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο να συνεισφέρει στις προσπάθειες των κρατών μελών και των εταίρων για να βελτιωθούν τα πράγματα και να επιτευχθούν οι στόχοι. Ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπορούσε ο σκιώδης εισηγητής μας να συμμετάσχει στις διαβουλές. Σας ευχαριστούμε. Δεμάτο παρακαλώ, σκιώδης εισηγήτρια, Δεμάτο. Και εγώ ευχαριστώ πρόεδρε τον ε, συνάδελφο για τη γνωμοδότησή του και σε ένα συγκεκριμένο εδάφιο ο συνάδελφος υπογραμμίζει ότι η Αρκτική θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας χώρος έρευνας ιδανικός για τον οικοτουρισμό, για την αηφόρο ανάπτυξη, νέες ενέργειες για το περιβάλλον και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που μπορούν να ε, ευημερούν με βάση καινοτόμα περιφερειακά τέτοια προγράμματα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την υψηλή οικολογική αξία αυτής της περιοχής ε, και για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής ε, από το 2014-2020 έχουμε θεματολογικά επιλέξει θέματα ε, και είναι πολύ σημαντικό τα λειτουργικά προγράμματα σε εθνικό και ε, υπερεθνικό επίπεδο να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα στοιχεία για μια πραγματικά αηφόρο ανάπτυξη που θα μπορεί να επιτευχθεί. Η τήξη των πάγων στην Αρκτική προέρχεται κυρίως από τις βιομηχανικές εκπομπές ρήπων της Ευρώπης και των ΗΠΑ και πρέπει εδώ να δούμε ότι ανεβαίνει επικίνδυνα το επίπεδο των θαλασσών. Πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη το θέμα που το οποίο αναφέρεται από μη κυβερνητική οργάνωση για τη δημιουργία ενός καταφυγίου στην Αρκτική όπου στην Αρκτική θα απαγορεύεται οποιαδήποτε εξορρυκτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους που να θέλουν να παρέμβουν από πλευράς μελών. Κύριε Νίλσον, εσείς θα θέλατε να απαντήσετε τώρα παρακαλώ. Α, Πρώτα να ακούσουμε όμως τους εκπροσώπους της Επιτροπής Περιφερικής Ανάπτυξης και μετά να τοποθετηθείτε. Σφάλμα μου αυτό, ζητώ συγγνώμη που το αγνόησα. Ο κύριος Γιωροσιέβιτς και ο εκπρόσωπος μετά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει τον λόγο λοιπόν να παρέμβετε. Σας ευχαριστώ από την Υπηρεσία ε, Εξωτερικής Δράσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη, διότι συνεργαζόμαστε από κοινού με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διατύπωση αυτής της κοινή ανακοίνωσης. Η ιδέα που είχαμε είναι, ήταν να τονίσουμε την επικοδομητική συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής. Γνωρίζουμε το γεωπολιτικό πλαίσιο βέβαια. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι στο περιφερειακό επίπεδο η συνεργασία μεταξύ των χωρών και με τη Ρωσία λειτουργεί και βαίνει καλώς. Και αυτό επίσης και από το Αρκτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα παρακολούθησα μια ad hoc συνεδρίαση σε σχέση με τους, τα, τις διαβουλεύσεις των ανώτερων αξιωματούχων ο Καναδάς, ε, η ΙΠΑ, η Ρωσία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία συνεργάζονται με εξαιρετικό τρόπο πολύ στενά και στρέφουν την προσοχή τους σε αυτά τα θέματα. Οι εντάσεις είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, δεν είναι υπαρκτές και υπάρχει και συνεργασία στην βόρεια διάσταση όσον αφορά το θέμα το προαναφέρθηκε. Αλλά έχουμε και το Συμβούλιο του, της θάλασσας του Μπάρεντς, το Συμβούλιο, Αρκτικό Συμβούλιο του Μπάρεντς, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ρωσία συνεργάζεται ε, και ενεργά έχουμε έναν αριθμό σχεδίων και πρωτοβουλειών διαμεθοριακής συνεργασίας και με την Ρωσία που λειτουργούν και εξελίσσονται. Η προσέγγιση είναι να κρατηθούν χαμηλή επίπεδα εντάσεων όσον αφορά τις δράσεις μας σε αυτή την περιοχή διότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα και υπάρχει και η βούληση να συνεργαστούμε. Και αυτό αντανακλά κιόλας και την ε, ευρωπαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας όσον αφορά για παράδειγμα την Αρκτική. Θα ήθελα να επανέλθω στην σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής περιφέρειας της Αρκτικής. Φυσικά η ανακοίνωσή μας προσπαθεί θέματα γύρω από τον Βόρειο Πόλο συνολικά σφαιρικά να τα καλύψει και να τα αντιμετωπίσει. Η Συμφωνία για την Αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλαγών των, των Παρισίων είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να καθοριστούν τα πλαίσια αυτών των δυνατοτήτων σε αυτό το πλαίσιο ώστε να συντονιστούν οι δραστηριότητές μας για την προαγωγή επενδύσεων σε αυτή την ευρύτερη περιοχή και ε, λειτουργούν τα πράγματα, προχωρούν και ε, θα έχουμε τον επόμενο Ιούνιο μια τέτοια εκδήλωση στη Φινλανδία που θα αποτελέσει πραγματικά ορόσημο για το βήμα το φόρουμ της Αρκτικής ε, για μας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα επίσης να πω ότι στο ίδιο επίπεδο σε αυτή την ανακοίνωση τοποθετούμε την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση και αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών και την άμβλυνσή τους, αποκινούμε προσπάθειες για την αηφορία, για την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτά συμπεριλαμβάνουν φυσικά και τη συνδρομή μας στους γηγενείς, στους αυτόχθονες λαούς. Και αυτά τα συνδυάζουμε και με τη διεθνή συνεργασία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πράγμα το οποίο και αυτό τονίζουμε και συνολικά στόχος αυτής της εργασίας για την Αρκτική είναι η υποστήριξη και της έρευνας και της καινοτομίας. Με υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας που είναι πολύ σημαντικές υποθέσεις και στη συνάντηση των αρμόδιων για τα θέματα της Αρκτικής το Σεπτέμβριο στην Ουάσιγκτον που διοργανώθηκε από τον Λευκό Οίκο τον, την Αμερικανική Προεδρία υπήρξε μια κοινή δήλωση για πρωτοβουλίες που υπεγράφει στη συνέχεια και συνεισέφερε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις διαβουλεύσεις και υπήρξαν σημεία που τονίστηκαν ότι με τον ορίζοντα 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, συνεισφέροντες όσον αφορά την έρευνα, την ε, επιστήμη, την ανάπτυξη και δίνουμε και σημαντικά κονδύλια για την έρευνα στην Αρκτική και αυτό δείχνει την εμβέλεια της συμμετοχής αυτής ε, ε, για τα θέματα Αρκτικής ε, στη διάσκεψη της Ουάσιγκτον. Ολοκλήρωσα εδώ, θα λάβει τον λόγο συνάδελφος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Γιώνα Κίλβα λέγομαι και είμαι στην Γαμαδέλτα Ρίτζιο. Τρία σημεία ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, σας ευχαριστώ όλους που αναγνωρίσατε την σημασία αυτής της συνεργασίας, της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ευχαριστώ που αναδεικνύετε και εσείς τη σημασία αυτής της συνεργασίας και θα υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρίτζια έχουμε 8 προγράμματα σημαντικά για την περιοχή, 2 ε, για την ε, Φιλανδία, 2 για την ε, Σουηδία και 4 διαπεριφερειακά, 2 διασυνοριακά, 2 διεθνικά. Πολύ αποτελεσματικά προγράμματα, λειτουργούν αίσια Ίσως διαβάσατε και την ανακοίνωση και είδατε ότι υπάρχει ένα διαπεριφερειακό ε, πρόγραμμα που αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα και λέμε ότι το ε, διαπεριφερειακό πρόγραμμα για την περιοχή της Αρκτικής ε, θα συγκροτήσει ένα δίκτυο αρμοδίων αρχών και εμπλεκομένων φορέων από επιμέρους περιφερειακά πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής. Επειδή είμαι αρμόδια για αυτό το πρόγραμμα, μπορώ να σας πω με χαρά ότι έχει αρχίσει ήδη ε, η συνεργασία, ε, δηλαδή συνεδριάζει η ομάδα εργασίας ε, και πρόκειται και για τα ΙΕΝΑΣ, e όχι μόνο για τα δικά μας προγράμματα, δηλαδή προγράμματα με τη Ρωσία, παραδείγματο χάρη. Αυτή, για αυτούς που ενδιαφέρονται έχω φέρει πολύ καλές εκθέσεις, πολύ ενδιαφέρουσες για να ξέρετε ε, τι γίνεται με τα πιλωτικά προγράμματα για να συγκεντρωθούν όλες οι χρηματοδοτικέ πηγές. Α, ευχαριστούμε. Ο κύριο Νίλσεν τώρα. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Παρατηρώ ότι μπορούμε σε πολλά σημεία να αναβαθμίσουμε αυτή την έκθεση, να βελτιώσουμε τη διατύπωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη. Χαίρομαι πολύ που ε, πολύ υποστηρίζετε τη διαπεριφερειακή συνεργασία σε αυτή την περιοχή. Ε, αυτό το δίκτυο των αεροκατοικημένων βορείων ε, περιοχών είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα προσφυλές συμμετείχα συγκεκριμένα και εγώ και νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ενισχύσει τη δράση σε αυτό το τομέα και τη συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα, διότι ε, πέρα από τις διαχειριστικές αρχές, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να μετάσχουν ε, ενεργά ε, στη διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων. Ε, τώρα δεν ξέρω αυτό που είπατε για τα εξωτερικά προγράμματα τις εξωτερικές υποθέσεις μάλλον μέσα σε αυτή την έκθεση. Ήθελα να σου πω μόνο ότι ε, είναι δύο οι συναρμόδιες επιτροπές ε, εξωτερικών υποθέσεων και περιβάλλοντος για να είμαστε αξιόπιστοι λοιπόν ας μην εκφραζόμαστε εμείς για ε, υποθέσεις ε, που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας μόνο τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς μας θα πρέπει να γύρουμε ε, για να έχουμε, παραμένουμε αξιόπιστοι και για να υπολογίζουν απόψή μας, νομίζω θα πρέπει να ε, περιοριστούμε στα ζητήματα αρμοδιότητάς μας. Έχω λοιπόν αυτή την αμφιβολία σε σχέση με την πρότασή σου, αλλά υπάρχουν πολλέ άλλε που μπορώ να ενσωματώσω και να βελτιώσω έτσι την ε, έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα Ολοκληρώνω τη συζήτηση. Θυμίζω μόνο πως η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι τη Δευτέρα 17 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Επόμενο σημείο. Παρουσίαση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή των επιδόσεων ε, τη πολιτική και τη συμμόρφωσης της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑΡΕΤΖΙΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μάρτιν. Θα έρθει στις 10 και 4 ο κύριος Μάρτιν, οπότε έχουμε 12-13 λεπτά, μπορούμε να πιούμε ένα καφεδάκι. 10 και 4 ξαναρχίζουμε, παρακαλώ.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

No,

Okay.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

και Αυτό μειώνει, Είναι το πω, να πόνεσμα, όλα αυτά. La mort, moi, ça, je Thank you.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

Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα εργασιών μας για σήμερα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Νίκλας Μάρτιν, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για την περιφερειακή πολιτική όσον αφορά την Γενική Διευθύνση Ρέγγιο για την περιφερειακή και πολιτική για τα αστικά κέντρα για τις πόλεις στις 14 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πακέτο προτάσεων Omnibus, προτάσεις που αφορούν την ενδιάμεση αναθεώρηση και όσον αφορά και την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Η πρόταση για την τροποποίηση αυτή και την προαγωγή αλλαγών για τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους για την χρήση αυτών των πλαισίων στήριξης. Ωστόσο, εμπεριέχονται και συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, ιδιαίτερα στο άρθρο 262 και εφεξής, που ξεπερνούν κατά πολύ τις εισαρθήσεις αλλαγές όσον αφορά το CPA και βασικές άλλες πράξεις. Και για αυτή την πρόταση από πλευράς του Κοινοβουλίου τώρα που βρισκόμαστε στην μέση ακριβώς, στην καρδιά των ευθυνών για αυτό το χαρτοφυλάκιο Υπήρξε μια αρχική συζήτηση στην Σύνοδο των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και στις 25 Οκτωβρίου θα επανεξεταστεί το θέμα, θα δοθεί συνέχεια. Είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση που θα παρουσιαστεί από εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διαμορφώσουμε εμείς την άποψή μας για αυτά τα θέματα. Έχετε λοιπόν τον λόγο κύριε Μάρτιν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να προσέλθω στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή σήμερα, να κάνω αυτή την παρουσίαση για αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η σωστή συγκυρία ως χρονική στιγμή για να το κάνω αυτό, για να σας δώσω συνολικά τις επεξηγήσεις για το γιατί προτείναμε και τι είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση να προσέρχομαι στη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτό που θα κάνω είναι θα επικεντρωθώ σε μία από τις αλλαγές όσον αφορά την πολιτική συνοχής, γιατί αυτά τα οποία προτείνονται θα έχουν επιπτώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής. Για να το εντάξω σε ένα συνολικό πλαίσιο, αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση αναθεώρηση και έτσι συνδέεται πάρα πολύ στα όσα ε, εκτίθενται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επικέντρωση στην ελαστικότητα, στην ευληγησία όσον αφορά τα νέα κονδύλια από πλευράς προϋπολογισμού. Τα κυριότερα σημεία εδώ είναι το τι μπορούμε δηλαδή να πράξουμε για την επιτάχυνση της υλοποίησης των διαθροτικών ε, και επενδυτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να απλουστεύσουμε αυτή την ε, υλοποίηση αυτών των δράσεων. Αυτά συνολικά είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως έχετε συνειδητοποιήσει είναι μια ευρεία δέσμη μέτρων, ε, η δέσμη Omnibus, με την ε, χρηματοοικονομική ρύθμιση και τους εξειδικευμένους κανόνες. Ήταν ε, επιλογή να το κάνουμε αυτό μέσα σε μια συνολική δέσμη μέτρων, διότι οι αλληλοσυνδεόμενες αλλαγές και σε σχέση και με τους κανόνες και κανονισμούς, αλλά και το κοινό θέμα της απλούστευσης και της στόχευσης, το καθιστούν αυτό αναγκαίο. Θα επικέντρω καθώς τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνδέονται ιδιαίτερα με την πολιτική συνοχή και τα ευρωπαϊκά επενδυτικά και ε, διαθωτικά ταμεία. Με τέσσερις άξονες θεματολογικά όπως και στην διαφάνεια αναφέρεται αυτό, δηλαδή μείωση του βάρους ε, για τους εμπλεκόμενους και όσους θα υποφεληθούν, συνέργεια των χρηματοοικονομικών μέσων και αύξηση δυνατοτήτων από πλευρά συνδυασμών των κρατών μελών. Κάποια νέα στοιχεία ε, θα δείτε και αρκετά σημαντικά στοιχεία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, το οποίο δεν υπήρχε όταν ε, είχαμε προχωρήσει, αλλά και στην ε, λεπτότερη ρύθμιση ε, και θα δείτε ύστερότερα ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις που θα μπορούσαν και μπορούν να διατυπωθούν με απλούστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη το έργο της υψηλής ομάδας αξιωματούχων με κάποιες συστάσεις που εξεπώνησαν και όλα αυτά εντάσσονται στην πρότασή μας και μια συγκεκριμένη ρύθμιση για το Ταμείο Αλληλεγγύης επίσης που θα αναφέρω στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το οποίο όλοι μας ε, έχουμε στην καρδιά μας ε, την ανάγκη να μειωθεί δηλαδή η επιβάρυνση για τους ε, όσους εποφελούνται για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εδώ οι κύριες αλλαγές αφορούν την απλούστευση όσον αφορά το κόστος όφελος πώς μπορούν οι εποφελούμενοι να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια χωρίς ε, να χρειάζεται να υπάρχει κάθε απόδειξη και εξόφληση για κάθε ευρώ που δαπανάτε. Το είχαμε αυτό υπόψη, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε στην πρότασή μας είναι ε, επεκτείνουμε αυτές τις προσπάθειες και τα, τις καθιστούμε πιο ειδικέ, δηλαδή για παράδειγμα αφαιρείται το άνω όριο για lump ε, που ήταν μία από τις επιλογές και υπήρχαν περιορισμοί. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που προξενούν κάποια συζήτηση. Είναι υποχρεωτική πλέον η χρήση της απλουστευμένης επιλογής ε, κόστους ωφέλους ε, και έτσι μειώνεται η επιβάρυνση για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να χρησιμοποιούν μία από τις απλουστευμένες επιλογές ε, για ποσά κάτω από 100.000 ευρώ. Και έτσι εντάξαμε στις γενικότερες προσπάθειες ε, το ETC έναν τρόπο υπολογισμού δηλαδή των άμεσων δαπανών και των δαπανών ε, στελέχωσης και αντίστροφα εντάσσουμε κάτι το οποίο εφαρμοζόταν μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δίνοντας τη δυνατότητα τα άλλα επιλέξιμα άμεσα ως δαπάνες ε, να μπορούν να ενταχθούν στους υπολογισμούς έχουμε και κάτι πιο καινοτόμο, πιο καινοτόμες δυνατότητες για την απλούστευση, για το κόστος ε, και για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας το σχέδιο προϋπολογισμού που είναι ένας προϋπολογισμός κομμένος και ραμμένος για τις λειτουργικές ανάγκες που θα μπορεί να λειτουργεί για όλα τα ταμεία και παίρνουμε και κάτι το οποίο βρίσκεται και στο δημοσιονομικό κανονισμό και θέτουμε αυτό στις κοινέ διατάξεις που το καθιστά δυνατό και εφικτό να δούμε πώς με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα συνδέεται η χρηματοδότηση. Τρόποι δηλαδή συνδυασμού των πληρωμών όσον αφορά τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Και τέλος δίνουμε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να δημιουργήσει ε, μία δυνατότητα ε, απλούστευσης ε, για τη διαμόρφωση του κόστους σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες με μεθοδολογία που καθορίζεται και με τον τρόπο αυτό η μεθοδολογία αυτή καθιστά βέβαια ότι θα μπορεί να γίνεται δεκτή Επίσης θα θυμόσαστε ότι μία από τις καινοτομίες που είχαμε στις κοινέ διατάξεις με τα κοινά σχέδια δράσης, joint action plans, για την ε, υλοποίηση μέρους προγράμματος ε, με βάση όρους, προϋποθέσεις ή επιδόσεις. Το πρόβλημα είναι ότι ήταν μια εξαιρετική ιδέα, αλλά κανένας δεν έδωσε συνέχεια σε αυτήν. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μια και δεν υπήρξε ενδιαφέρον, θα έπρεπε να γίνουν σαφώς κάποιες αλλαγές για να γίνει πιο ε, φιλικό προς τους χρήστες αυτό το εργαλείο. Διότι είναι σημαντική λιθος η δοκιμασία για ένα διαφορετικό τρόπο για τις επιδόσεις ε, και την αξιολόγησή τους. Το διευκολύναμε λοιπόν ε, σε σχέση με τα ανώφλια όσον αφορά την ελάχιστη ε, κοινή δαπάνη ή την επιμεριζόμενη κοινή δαπάνη και ε, σε σχέση με τα πιλωτικά προτείναμε για το πρώτο κοινό σχέδιο δράσης δεν θα υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει ή προδιαγραφές και σε μικρή κλίμακα θα μπορεί να λειτουργήσει και όσον αφορά το περιεχόμενο και τις απαιτήσει είπαμε ότι δεν χρειάζεται διαφορετική ξεχωριστή διαχειριστική επιτροπή Επιτροπή, αλλά μπορεί η Εποπτική Επιτροπή να χρησιμοποιείται. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν τα οποία απλουστεύουν εντασσόμενα στις διαδικασίες, στις ε, διεργασίες αυτές και θα τα καταστήσουν όλα αυτά πιο ελκυστικά και όταν θα υπάρξουν, θα ε, έχουν παγιωθεί αυτές οι αλλαγές θα δοκιμάσουμε όλα αυτά πιλωτικά με τα κράτη-μέλη διότι θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ένα χρήσιμο πρότυπο αυτό για την περίοδο και μετά το 2020 και χρειάζεται και πρακτική εμπειρία και πρακτική και πείρα που πρέπει να συλλεγεί πρώτα. Αυτά σε σχέση με το πρώτο τμήμα όσον αφορά την μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά την βελτίωση των συνεργειών. Και αυτό πάλι είναι κάτι που γνωρίζω ότι γι' αυτό, ε, σε αυτό επικεντρώθηκε ιδιαίτερα η δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και το εξετάσαμε σε διαφορετικούς τομείς όσον αφορά τον ορίζοντα 2020. τα οποία προέκυψαν περίπου πριν από ένα χρόνο και ένα από τα ζητήματα που υπογραμμίστηκε είναι η ανάγκη του να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει υψηλού επίπεδου συμπληρωματικότητα μεταξύ των ε, πόρων ΕΣΥ και αυτών του νέου μέσου, το οποίο διαχειρίζεται η IB, η Τράπεζα των Επενδύσεων. Και καθότι δεν το γνωρίζαμε αυτό, δεν μπορέσαμε να εντάξουμε τα στοιχεία που θα επέτρεπαν μια καλή διάρθρωση μεταξύ των δύο μέσων. Εκδώσαμε ένα εγχειρίδιο που εξηγεί πώς αυτό μπορεί να γίνει, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει η επιθυμία αυτό να απλουστευθεί και να διευκολυνθεί. Και αμέσως μετά θα εξηγήσω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Σε διαφορετική κλίμακα, τελειοποιήσαμε το σχέδιο που είχαμε επί της διατάξεως που λέει ότι η ίδια επιχείρηση, το ίδιο έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από διαφορετικές πηγές. Το οποίο επιτρέπει στα, στους πόρους ΕΣΥ να συνεργαστούν με τους πόρους του ορίζοντα 2020 μεταξύ άλλων. Ένα από τα ζητήματα ήταν ο έλεγχος σχετικά με τις δαπάνες που απλουστεύτηκε διότι μπορεί να γίνει προράτα πλέον. Δηλαδή το 70% της ε, δραστηριότητας ε, θα χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα με πόρους ε, περιφερειακής ανάπτυξης και το υπολοιπόμενο 30% από άλλο πρόγραμμα ή από άλλο ταμείο, όπως ορίζοντας 2020 για τα ερευνητικά. Πρόκειται λοιπόν για μια ρύθμιση, αν θέλετε, μια διευκόλυνση. Ας πάμε τώρα στις λεπτομέρειες του συνδυασμού των με τα έύση. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή παραδοσιακή θα λέγαμε επιλογή, όπου η διαχειριστική αρχή διαχειρίζεται πόρους ESIF και το συνδυάζει με επενδύσεις ΕΦΣΥ επί τη βάση των συζητήσεων που είχαμε με την Τράπεζα Επενδύσεων. Προτείνεται λοιπόν ότι ο συνδυασμό αυτός εκινεί μια νέα δέσμη διατάξεων σε συγκεκριμένο άρθρο, νέο άρθρο, σχετικά με δημοσιονομικά μέσα που θα διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις που θα διευκολύνουν ακριβώς το συνδυασμό των δύο μέσων. Προκειμένου τώρα να έχουμε κάποιες εγγυήσει για τη χρησιμοποίηση των πόρων ΕΣΥ, έχουμε ένα μέγιστο όριο συμμετοχής. Θέλουμε δηλαδή να εξασφαλίζουμε ότι όταν εισέρχονται, εισραίουν οι πόροι ΕΣΥ, θα πρέπει να έχει υπολογιστεί η πρώτη απώλεια στο δημοσιονομικό μέσο. Δηλαδή λέμε ότι δεν πρέπει να είναι άνω, άνω του 25% του συνόλου. Με μεγαλύτερη ευελιξία όμως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Και έχουμε ένα, μια άλλη δέσμη κανόνων που διευκολύνει ώστε να έχουμε ενιαίο σετ κανόνων για να έχουμε και τους δύο κανόνες από κοινού. Απλουστεύει λοιπόν την εξάντια αξιολόγηση διευκολύνει και απλουστεύει την υποβολή εκθέσεων, επιτρέπει 100% χρηματοδότηση και σημαίνει επίσης ότι η διαχειριστική αρχή μπορεί στα πλαίσια επενδυτικής πλατφόρμας να χρησιμοποιήσει τους πόρους εύση κτλ. Έχουμε δηλαδή αν θέλετε ένα ενιαίο σημείο αναφορά σχετικά με τις εφαρμοστές διατάξεις. Επίσης, καθότι το ΕΦΣΙ είναι ένα νέο μέσο υβριδικό θα έλεγε κανείς μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όταν η Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει κανονικά, αυτό λογίζεται ως ιδιωτική εισφορά. Ιδιωτική πόρη. Όταν όμως χρησιμοποιούνται πόροι ΕΣΥ ή ΕΣΑΙ, αυτό είναι δημόσια εισφορά. Το ΕΦΣΙ είναι ανάμεσα στα δύο. Διότι υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και θεωρείται δημόσια εισφορά, αλλά, αλλά προέρχεται από την Τράπεζα Επενδύσεων όπως και άλλες επενδύσεις. Επομένως είχαμε ένα κενό, για να το πούμε έτσι, σχετικά με το πώς θα έπρεπε να διαχειριστούμε όλα αυτά, γιατί σε κάποια διαρθρωμένα χρηματοοικονομικό, χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει κανείς να επιτρέψει διαφοροποιημένη διαχείριση συγκεκριμένων επενδυτών. Συντάξαμε λοιπόν τη διάταξη του άρθρου ώστε να είμαστε συγκεκριμένοι και σαφείς σχετικά με τους πόρους που θα προέρχονται από το ΕΦΣΙ και επομένως διευκρινίζεται πλέον λεπτομερώς η δυνατότητα της χρησιμοποιήση των πόρων ΕΦΣΙ ως εκείνη που θα καλύπτει την μικρότερη συνεισφορά καταβολής ή την πρώτη απώλεια συγκεκριμένου προγράμματος ή έργου. ώστε να μην εστιαστούμε μόνο στις περιφέρειες, στις περιφέρειες εκείνες όπου το ποσοστό κινδύνου είναι, αν θέλετε, πιο εύκολο προς διαχείριση ή μικρότερο. Αυτά είναι τα σχετικά με την ε, νομική αποσαφήνιση που χρειάζεται, τις διευκρινίσεις τις νομικές και τεχνικές που χρειάζονται ώστε να συμμετάσχουν οι επενδυτές. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη επιλογή. Λόγω του νέου άρθρου 125 στο δημοσιονομικό κανονισμό, που έχει δύο στοιχεία που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τμήμα των πόρων που δικαιούται από το ΕΣΥΦ ώστε να αντισταθμίσει τη δυνατότητα κινδύνου. Είναι δυνατότητα δηλαδή για ένα κράτος μέλος να κάνει μια αίτηση να μεταφερθούν τμήματα των πόρων έσυφ στα οποία έχει δικαίωμα προς τον προϋπολογισμό ώστε να υποστηρίξει από εκεί τους πόρους εύση και έτσι να αυξήσει την επενδυτική ικανότητα της τράπεζας. Και επομένως η πίστοση αυτή αφαιρείται από τους πόρους ESI και η αύξηση επενδυτική ικανότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να είναι πλέον τμήμα τη κανονική αν θέλετε δημοσιονομική διαδικασία. και προκειμένου το 125 να λειτουργεί στην πράξη προτείναμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του κανονισμού ώστε τα κράτη-μέλη μέχρι συγκεκριμένη προθεσμία να μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν τη διάταξη αυτή. Αυτά φυσικά για μελλοντικέ για, μελλοντικ, για μελλοντικούς προϋπολογισμούς. Τώρα θα θυμάστε επίσης ότι είχαμε συγκεκριμένες διατάξεις στον κανονισμό για χρηματοδοτικά μέσα ώστε να έχουμε ένα μια πλήρη δέσμη διατάξεων ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε την αυξημένη χρήση των μέσων προς την οποία να αποσκοπούσαμε. Θέλαμε δηλαδή να επιτρέψουμε μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Και η πρώτη ουσιαστική αλλαγή είναι η επιλογή των διαχειριστών των ταμείων. Πρόκειται για υπηρεσία και επομένως καλύπτεται από την οδηγία δομησίων προμηθειών, πρέπει να περάσει κανείς από τη διαδικασία του διαγωνισμού κτλ. Οι υφιστάμενες εξαιρέσεις είναι για την Τράπεζα Επενδύσεων και το EIF, λόγω διατάξεων συνθήκης. Αυτό το που προτείνουμε τώρα είναι άμεση, άμεσο ορισμό που μπορεί να γίνει από κράτος μέλος για το διαχειριστή, ώστε εθνικές τράπεζες προώθησης να αναλάβουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες ένα τμήμα το οποίο θα διαχειρίζεται η Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό συζητήθηκε στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση και το είχαν ζητήσει διάφορα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι αυτό θα απλουστεύσει τη διαχείριση των δημοσιονομικών μέσων και την άμεση ανάθεση, την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένες τράπεζες εθνικές επενδυτικές εν πάση περιπτώσει που θα έχουν σχηματιστεί για αυτό το σκοπό. Επίσης είχε σημειωθεί μια άμεση ανάγκη να, να υπάρξει ρευστότητα για τις επιχειρήσεις. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε κάπως καθυστερημένα, διότι είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις από τα κράτη-μέλη και ήρθε κάπως αργά, αλλά έχουμε πέντε κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτή την πρωτοβουλία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προτείνεται η επέκταση μέχρι το τέλος περίοδου για τη δυνατότητα χρησιμοποίηση του μέσου αυτού, της πρωτοβουλίας αυτής. Είναι άλλο λοιπόν ένα μέσο που είναι διαθέσιμο για τα κράτη-μέλη προκειμένου να στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και κάποια άλλα τεχνικά στοιχεία, μικροδιορθώσεις και βελτιώσεις εκεί που θέλαμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα κάποιων διατάξεων για ε, τον έλεγχο των IFI και της ε, Τράπεζας Επενδύσεων προτείνουμε μια διαδικασία υποβολής εκθέσεων για τα κράτη-μέλη που προέρχεται από τους ελεγκτές της Τράπεζας Επενδύσεων ώστε να αποφεύγουμε επικάλυψη του, της όλης διαδικασίας της ελεγκτικής. Με δημοσιονομικές ε, διορθώσεις όπου αν υπάρχει συγκεκριμένη απόκληση δεν θα οδηγεί σε αναθεώρηση του όλου μέσου. Επίσης λάβαμε υπόψη και τα αρνητικά επιτόκια που πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν, αν θέλετε, μια πραγματικότητα. Τώρα λάβαμε και αυτό υπόψη και το συνυπολογίζουμε. Συνολικά, επομένως, από όλες τις τροποποιήσεις στο CPR, Έχουμε το αποσταμένο κόστος αφενός και το άλλο για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Και προχωρώ στην τρίτη θεματική, αν θέλετε, την ευελιξία. Εδώ ε, ε, προσθέσαμε συγκεκριμένη διάταξη που λέει ότι για όλα τα ταμεία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υποστηρίζονται δαπάνες που είναι σχετισμένες με την μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό αποτυπώνεται και στον ε, κανονισμό EIDF. Διευκολύνουμε τις διαδικασίες σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις, γιατί θέλουμε αυτό το κείμενο να είναι ζωντανό, να επικαιροποιείται διαρκώς. Υπήρξαν κάποιες σάφειες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να γίνονται για αυτό, το κάναμε η μεσαία τελεία είναι για το άρθρο 125 του Δημοσιονομικού. Και για το ΕΦΣΙ υπάρχει μια γενική δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων από τα ESI προς, όπως έλεγα, τον ενωσιακό προπολογισμό για να χρησιμοποιηθεί για άλλα μέση. Επομένως, στο CPR εντάξαμε μια διάταξη που καθιστά δυνατό για κράτος μέλος να μεταφέρει ένα τμήμα της πίστοσης του εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ιδανικά εντός της προγραμματικής περίοδου προς τον υπολογισμό ώστε να υποστηριχθούν π.χ. διαδικασίες έρευνας στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Επίσης, κάποιες ε, τροποποίησεις που προτείναμε για τον κανονισμό ERDF ε σχετικά, όπως έλεγα, με τη δυνατότητα της υποστήριξης επενδύσεων που θα σχετίζονται με την μετανάστευση και το άσυλο και τις πρόσφυγες. Υπάρχει μία προτεραιότητα που καλύπτει την ε, ε, υποδοχή και την ένταξή τους και παρέχει κάποια σαφήνεια σχετικά με τους πόρους που χρησιμοποιούνται, τις δαπάνες δηλαδή που γίνονται σχετικά με αυτά. Παρέχεται δηλαδή ένα σαφέστερο πλαίσιο και αποφεύγονται κάποιες νομικές αμφιβολίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογή. Έχουμε επίσης δείκτες πεδίου εφαρμογή σχετικά με την χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών και άλλο σημείο που είχε τεθεί από διάφορα κράτη-μέλη, περιορισμός για τη χρησιμοποίηση υποδομών ε, σε περιπτώσεις ε, τουριστικών και πολιτιστικών επενδύσεων ε, κάποια κράτη-μέλη θεώρησαν ότι αυτό ήταν προβληματικό, δεν ήταν σαφές τι εννοούσε και ήταν υπερβολικά περιοριστικό. Επομένως αφαιρέσαμε διαγράφει η μικρή κλίμακα του μέσου εκείνου, της διάταξης εκείνης. Επίσης εισήχθη μια ευελιξία ε, σχετικά με τις ε, δράσεις που οδηγούν σε πρόσθετα έσοδα ώστε να μπορούν τα κρατημέλη να ορίζουν τις δικές τους καταποκοπήν καταβολές, ιδιαίτερα σε εθνικούς τομείς όπου είναι πολύ δύσκολο εμείς να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή να το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα και ενώ ένα κράτος μέλος μπορεί να, να έχοντας τα στοιχεία που χρειάζονται να ορίσει τις ε, καταβολές καταποκοπήν με τις απαραίτητες ε, ε, αφαιρέσεις ποσών που πρέπει να γίνουν εσόδων. Άλλο ένα στοιχείο για τα έργα μεγάλου ενδιαφέροντος. Έχουμε ένα fast track, δηλαδή μια επιταχυμένη διαδικασία μέσω ανεξάρτητης ε, αναθεώρησης ποιότητας ώστε να επιταχύνει τη διαχείρισή τους, αλλά δεν είχαν κίνητρα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το fast track αυτό, γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δαπάνες εντός του δελτίου μετά τη λήψη της απόφασης Κομισιόν. Και επομένως, αφαιρέσαμε αυτό το αντικίνητρο, αν θέλετε. Και μόνο κάποιες ακόμα τροποποίησεις που έγιναν υπό το fine tuning, διευθυνίζοντας κάποιες δυσκολίες που υπήρχαν για τον ορισμό των φυσικών προσώπων, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, των ενδιαμέσων σωμάτων ή φορέων, των ε, Συμβουλίων Ανάπτυξης και ITI και επίσης της στήρησης εγγράφων δίνεται η δυνατότητα να τηρούνται ηλεκτρονικά, αλλά υπήρχαν διατυπώσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη ε, με συγχωρείτε σχετικά με τη διατύπωση του κειμένου εκεί, τεχνική βοήθεια επίση. αυξημένη ευελιξία για τη χρησιμοποίηση τη τεχνική αρρωγή και των ανωτάτων ορίων, Δεφνίζοντα ότι για τα πράγματα ETC η ίδια αρχή πιστοποίηση και αρχή διαχείριση, μάλλον η διαχείριση και η πιστοποίηση μπορεί να γίνει υπό τον ίδιο φορέα. Και κάποιες ε, διασταυρούμενες ε, παραπομπές. Και στον κανονισμό ECF χρειαζόταν κάποια τακτοποίηση. Οι διατάξει απλουστευμένου κόστου ε, ομαδοποιήθηκαν αν θέλετε και ξεκαθαρίσαμε κάπως και τους δείκτες. Και είχα αναφέρει από την αρχή για κάποιες αλλαγές στο Ταμείο Αλληλεγγύης, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε προϋπολογισμό. Είχαμε μία προβολή, αν θέλετε, και κάθε φορά που χρειαζόταν να αντλήσουμε από το Ταμείο, τροποποιούσαμε τον κανονισμό, τον προσωρινό κανονισμό. Τώρα προβλέπεται συγκεκριμένη συγκεκριμένο κονδύλι του προπολογισμού, το οποίο θα μπορεί να κινητοποιείται. Αυτό δεν επηρεάζει διαδικασία ω προ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που ούτω ή άλλω πρέπει να εγκρίνουν την άγκληση ή την κινητοποίηση των πόρων κάθε φορά. Αυτά ε, ολοκληρώνουν την συνοπτική παρουσίαση των ε, τροποποιήσεων. Προσπάθησα να διαφοροποιήσω μεταξύ μεταξύ κάποιων πιο ουσιαστικών και κάποιων πιο τεχνικών τροποποίησεων, αλλά όλες αποσκοπούν στην απλούστευση και τη βελτίωση του ε, νομοθετικού πλαισίου. Αυτό που είναι σημαντικό πλέον είναι η όλη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της συζήτησης που θα οδηγήσει στην έγκριση των τροποποίησεων αυτών να λύσει όσο πιο ομαλά γίνεται διότι ο σκοπός είναι να έχουν θετική επιρροή από των προγραμμάτων ε, μέχρι το 2020. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Μάρτιν. Ήταν ε, περιστατωμένη και ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Βλέπουμε πόσο περίπλοκες είναι οι προτινόμενες αλλαγές μέσα από την παρουσίασή σας. Δύσκολα ε, έχει κανείς μια γενική άποψη των αλλαγών ε, στις επιμέρους λόγω της περιπλοκότητας της πρότασης. Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα θα αρχίσει η συζήτηση. Η κυρία Κρέα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτιν, για τα όσα μας εκθέσατε τουλάχιστον για την αρχική κατάσταση φωτίζει η παρέμβασή σας κάποια πράγματα, τα αποσαφηνίζει. Αυτά τα οποία μας εκθέσατε σε μια πρώτη αντίδραση μπορώ όλα να τα τονίσω και να τα δεχτώ. Θα έδιναν όλα αυτά την δυνατότητα να πετύχουμε απλουστεύσεις και μείωση της γραφειοκρατίας χωρίς αμφιβολία και το δυνατόν γοργότερα θα πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά σίγουρα μόνο που ειλικρινά δεν κουράζομαι να επεξηγώ αυτό το οποίο βρίσκω αξιοπερίεργο το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια διαδικασία την παρουσιάζει ως omnibus διαδικασία σφαιρική και συνολική. Φυσικά υπάρχει διασύνδεση στο δημοσιονομικό κανονισμό του σώματος. Ωστόσο όλα αυτά τα οποία προτείνονται ως αλλαγές θίγουν σε βάθος ε, την ουσία της πολιτικής σύνοχης και δεν αφορούν μόνο την απλούστευση γενικά ή γενικότερα, αλλά αφορούν ε, ουσιώδη τμήματα της πολιτικής που αλλοιώνονται για την πολιτική σύνοχη. Δεν αμφιβάλλω ότι θα σας υποστηρίξει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την πολιτική σύνοχη για τα προγράμματα για πρόσφυγες ε, και ετούντες άσυλο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, θα σας υποστηρίξει το Ευρωκοινοβούλιο. Πρόκειται όμως για σε βάθος αλλαγές της ουσίας της πολιτικής συνοχής και στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων για την αποκλειστική αρμοδιότητα που θα έπρεπε να εξεταστεί επιμέρους το θέμα. Ή να πάρω ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάμαι πολύ καλά τις έντονες αντιπαραθέσεις και συζητήσεις μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου και για τα θέματα επίσης ποια κονδύλια θα εγγράψουμε όσον αφορά τα πολιτισμικά μνημεία, τα μνημεία πολιτισμού. Ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με υποστήριξη του Κοινοβουλίου με απόλυτη σαφήνεια να καθοριστεί ότι δεν θα έχουμε ένα τεράστιο ποσό συλλήβδιν και ισοπεδωτικά απλά και μόνο για μουσεία ιστορικά και άλλα, αλλά ότι θα θέλαμε όταν αυτά τα κονδύλια θα διατίθενται να χρησιμοποιούνται με πιο ζωντανό και έντονο τρόπο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για τη δημιουργία αεφόρου ανάπτυξης. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί φυσικά να έχει αλλάξει την άποψή του σήμερα. Δεν το αμφισβητώ αυτό, δεν προδικάζω πώς θα αποφασίσουμε, αλλά είναι μια απόφαση που εδώ στην Περιφερειακή Επιτροπή πρέπει να ληφθεί υπόψη και να προετοιμαστεί και με τα κράτη-μέλη σε τριμερή διάλογο να μπορέσει να συνεξεταστεί. Και στην διαδικασία όμνιμπους που προτείνετε εσείς δεν είναι δεδομένο αυτό, δεν διασφαλίζεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας στη συνάντηση συνάντηση συντονιστών που θα προετοιμάσουμε για απόφαση αυτά τα θέματα θα το συζητήσουμε αυτό. Είναι αδιανόητο για μας και ασύλληπτο υπό το πλαίσιο για παράδειγμα της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών ή Ελέγχου Προϋπολογισμών προϋπολογισμού να γίνει η δουλειά από αυτούς ε, όταν έχουμε μια τόσο στενή διασύνδεση που θα πρέπει και υπό δική μας αρμοδιότητα να εξεταστεί το θέμα. Γιατί διαφορετικά στον ε, τριμερή διάλογο λόγο οι, αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει και με τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να διαπραγματευτούν αυτά τα θέματα. Και δεν πιστεύω ότι σε σχέση με την επιβράδυνση των διαδικασιών αυτό θα προξενήσει κάποια επιβράδυνση όταν εμπλακούμε εμείς. Η Περιφερειακή Επιτροπή το έχει αποδείξει ότι επανειλημμένα μπορεί πολύ αποτελεσματικά να εργάζεται και να διαπραγματεύεται επ' αυτών των θεμάτων. Και πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή προϋπόθεση αυτή, ώστε οι διαδικασίες να μπορέσουν γοργά να ολοκληρωθούν. Η άποψη ότι σε μια μεγάλη διεργασία όμνιμπους σφαιρικά μπορούν όλα να καλυφθούν, πρέπει να εξεταστεί αυτό ιδιαίτερα προσεκτικά. Αν μία μόνο κοινοβουλευτική επιτροπή αναχαιτήσει ή τροχοπεδίσει τα πράγματα, τότε παγώνουν όλα και δεν θα προχωρήσει τίποτα. Και μπορεί σε ένα σημείο κάπως ε, περισσότερο να διαρκέσουν τα πράγματα ή να καθυστερήσουν λίγο περισσότερο αν εμπλέκονται όλοι όπως πρέπει. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει όμως τροχοπαίδηση συλλήβδιν, συνολική. Είναι πράγματα αυτά που πρέπει νομίζω να τα θα δούμε και που μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, προτάσεις ε, επιμέρους που έχουν διατυπωθεί. Ίσως να διατυπώσω μήπως αυτή την ανεδή κάπως ερώτηση προς εμάς. Το είπα κάπως ε, χαλαρά. Δεν είναι δυνατόν σε σχέση με την πολιτική συνοχή να αποσυνδεθούν τα πράγματα σε σχέση με τη διασύνδεσή τους με το σχέδιο, με το πρόγραμμα Juncker. Υπήρξε αυτή η δέσμευση, η υπόσχεση από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι δικές του απόψεις ε, για αυτό το, ε, για αυτό το ποσό που θα διατεθεί θα δημιουργήσουν μοχλευτική ε, επενέργεια που θα μπορέσει να δράσει θετικά. Αν τώρα όχι μόνο κάποια ιδιωτικά κονδύλια αλλά de facto η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με κρατικά και δημόσια κονδύλια για τη συγχρηματοδότηση θα συνεμπλέκεται δεν είναι αυτή η αρχική επιλογή που είχαμε επιλέξει και πείτε μου σας παρακαλώ λοιπόν πώς πρακτικά με τις δικές σας προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προλιάνετε το έδαφος για να γίνει κάτι τέτοιο ή μήπως θα υπάρξουν επιπρόσθετες ε, ε, επιπτώσεις από τις, από τις συνέργειες. Αυτό θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νοβάκοφ παρακαλώ. Επόμενος αγώνα. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή μου, διότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για την ε, απλοποίηση του συστήματος και διαπιστώνω ότι ένα χρόνο μετά έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένα βήματα για το μέλλον. Σίγουρα ε, θα περιμένουν ε, πληθώρα ερωτήσεων οι εκπρόσωποι της Επιτροπής από πλευράς μας. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το εξής. Πώς ε, θα οργανωθούν οι εργασίες γενικότερα και ειδικότερα στο Συμβούλιο. Διότι είναι 15 οι κανονισμοί και τα άρθρα. Είναι εκατοντάδες σελίδες ε, τροπολογίες, είναι ε, θα, ε, μεγάλος φόρτος εργασίας που μας περιμένει. Θα υποδιαιρέσετε ίσως σε τμήματα την πρότασή σας για λόγους πραγματογνωμοσύνης, διότι υπάρχουν τροπολογίες που είναι λίγο ασύνδετες με το ζήτημα. Όταν μιλάμε για την περιφερειακή ανάπτυξη, και τα διάφορα ταμεία και θα υποστηρίξω την κυρία Κρέολ για τους ε, πρόσφυγες. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πότε ακριβώς και θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα το χειριστούμε και με ποιες διαδικασίες θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και διαφανείς, ε, κυρίως στη σχέση με τους πολίτες. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό. Πώς ακριβώς έχετε ε, προγραμματίσει το χρονοδιάγραμμα. Είναι πρόωρο τώρα να μιλήσουμε για συγκεκριμένε ημερομηνίε. Τα αναγνωρίζω όμως καλό θα ήταν ε, να έχουμε μια προοπτική για να ξέρουμε τι θα περιμένουμε. Α, και για κάποιες άλλες προτάσεις. Ξέρω πόσο ε, δύσκολο περίπλοκο ζήτημα είναι η απλούστευση ακόμη και όταν μιλάμε για διοργανική συνεργασία. Η υψηλή ομάδα εργασίας έχει 12 ε, λέξεις στον τίτλο του. Αυτό είναι δηλαδή ο φορέας που θα χειρίζεται την απλούστευση και έχει 12 ε, λέξεις στον τίτλο του. Αυτό το ε, σώμα, αυτή η επιτροπή. το λέω έτσι για να καταδείξω την περιπλοκότητα του ζητήματος Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μία ταξινόμηση και πέρα από το feedback από εσάς να έχουμε και feedback από τους δικαιούχους ούτως ώστε να έχουμε αυτό το πίνακα βαθμολογίας επιδόσεων από, και από τους δικαιούχους. αν ο έλεγχος που γίνεται στους δικαιούχους βασίζεται στον κίνδυνο, όσοι έχουν καλές επιδόσεις να ελέγχονται λιγότερο. Και όσοι ε, παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο λάθος, δεν λέω απάτη, λάθος, θα μπορούσαν ενδεχομένω να υπάρχουν σε αυξημένους ελέγχους. Νομίζω αυτό θα βοηθούσε. Και έτσι θα μειωθεί και το άκθος που φέρουν οι δικαιούχοι. Τέλος. Μιλάμε για την απλοποίηση του συστήματος ε, και αυτό το είδους η τροποποίηση του νομικού πλαισίου με διάφορους τρόπους μας αφήνουμε το εξής ερωτηματικό. Αυτός είναι ένας οδικός χάρτης ε, σε σχέση με την εφαρμογή των ε, αλλαγών στα κράτη-μέλη. Το συζητάμε τώρα και τι εννοώ. Με κάποιο τρόπο θα εγκριθούν οι αλλαγέ. Πώς θα γίνει όμως να δούμε με το ποιο τρόπο εφαρμόζονται ε, στα κράτη-μέλη, Πώ επηρεάζονται οι δικαιούχοι, η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που θα εφαρμόσουν τις αλλαγέ. Είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε. Μαλέτητς. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση, για τις προτινόμενες αλλαγές είναι κοινό ο στόχο και είναι ευπρόσδεκτε οι αλλαγέ. Θέλουμε να ε, επισπεύσουμε την εφαρμογή ε, των ε, την απορρόφηση των κονδυλίων των ταμείων στα κράτη-μέλη και για να γίνει αυτό όντως πρέπει να απλοποιήσουμε τους κανόνες. Με όλες αυτές τις αλλαγές όμως αναρωτιέμαι, όντως θα επισπεύσουμε την υλοποίηση Και η Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για να γίνουν πιο εφαρμόσιμοι οι κανόνες. Με ποιο τρόπο θα συνεργαστείτε στενότερα με τα κράτη-μέλη για να επιτύχουμε ουσιαστική υλοποίηση. Αυτό το SEO, πολύ μου αρέσει, το Simplified Cost Option, λέτε θα είναι υποχρεωτικό. Εξαιρετική ιδέα. Πού θα τραβήξουμε τη γραμμή σε σχέση με αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν. Πολλοί δεν τη χρησιμοποιούσαν αυτή την αλλακτική λύση, η SEO. Για ποιο λόγο. Εμένα προσωπικά μου είπανε αν εστιάζονταν μόνο στο SEO είχαν προβλήματα με τους ελέγχους, και ε, τους οικονομικούς ελέγχους και δεν εστιάζονταν ε, στα αποτελέσματα αλλά στο input. Και αυτό είναι τελείως αντικρουόμενο στόχος ε, Γι' αυτό και χρειάζεται γενικότερη αναβάθμιση του συστήματος για να μπορέσουν να είναι εφαρμόσιμες αλλαγές. Γι' αυτό υποβάλλω την ερώτηση. Τη συνέργειας. επίσης, πολύ καλή ιδέα για το συνδυασμό διαφόρων ταμείων. Είχαμε πάρα πολλές ομάδες εργασίες και ακροάσεις για αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο για τις συνέργειες και ιδίω ανάμεσα στα ταμεία ΕΣΥ και τον ορίζοντα και ε, είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις διαφορές στους κανόνες. Στον ορίζοντα έχουν διαφορετικούς κανόνες για τις κρατικές προμήθειες, ε, για τους ελέγχους ε, κατά τη διαστολή με το, τα ταμεία ΕΣΥ και δύσκολα συνδυάζονται βεβαίως. Είπατε στη διάρκεια της παρουσίασής σας ότι με ποιο τρόπο ε, σκοπεύετε να εφαρμόσετε όλους αυτούς τους κανόνες με στόχο την πρόθεση της καλύτερης εφαρμογής στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε, Δεμάτο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσία του εδώ και που μας εξήγησε τη δουλειά αυτή. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω περισσότερες ε, διευθυνήσεις, ιδιαίτερα επί της συνέργειας μεταξύ των ΕΣΥΦ και του ΕΦΣΥ. Εμείς έχουμε μεγάλες απορίες, τις είχαμε εκφράσει και για την προστιθέμενη αξία του ΕΦΣΥ, διότι τα μεγέθη αυτά βασίζονται επί προβολών, όχι επί εγγυήσεων για τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνουμε ότι πρακτικά ε, το ε, ΕΦΣΥ ενεκρίθη μετά το CPR και δεν φτάνουν απλές κατευθύνες γραμμές, αλλά δεν σας φαίνεται κάπως επικίνδυνο να προτείνουμε τροπολογίες στον κανονισμό ναι. που υποτίθεται ότι ε, ενισχύουν τη συμπληρωματικότητα των δύο μέσων αλλά που δεν διέπονται τη διαφάνεια σχετικά με τα κονδύλια που έχουν, που έχουν καταχωριστεί σε, σχέση με συγκεκριμένα προγράμματα. Επίσης, η προτεραιότητα σχετικά με τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου ε, λέτε ότι αυτό γίνεται για να απλωστευθούν τα έργα και τα προγράμματα που αφορούν στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αλλά ε, εγώ προερχόμενοι από μια χώρα η οποία αποδέχθηκε πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες ε, περιφέρειες ε, του δικού μας νότου ή περιφέρειες της Ελλάδος που αντιμετωπίζουν σημαντικότατη πίεση λόγω της κρίσεως και που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική συνοχή για να αντισταθμίσουν τα προβλήματα αυτά, να τα αντιμετωπίσουν. Και δεν είναι μόνο ε, πρόβλημα των ε, περιφερειών αυτών, είναι πρόβλημα της, ε, όλης της Ευρώπης. Μου φαίνεται κάπως επικίνδυνο για τις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν πως, δηλαδή κονδύλια προερχόμενα από τέτοια μέσα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στάει κάποιο άλλο το λόγο. Για παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ενστάσεις, ο κύριος Μάρτιν, λοιπόν, ήρθε η ώρα των απαντήσεων. Σας ευχαριστώ. Πολύ ευστόχες οι ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Να αρχίσω με τα πιο θεσμικά ζητήματα. Γιατί τα συγχωνεύσαμε όλα σε ένα πακέτο και ποιο, ποιες επιπτώσεις έχει αυτή η επιλογή. Η Επιτροπή παρουσιάζει αυτό το πακέτο στα πλαίσια της, ε, των προτάσεων ενδιάμεσης αναθεώρησης. Νομίζω ότι στην ανακοίνωση εξηγείται με σαφήνεια ε, για ποιο λόγο το κάναμε αυτό. Ίσως καλό θα ήταν να έχουμε κατά νου πως... Ε, ίσως... Από τους κινδύνους που επολοχεύουν ε, είναι και αυτό φαίνεται σε συζητήσεις ε, και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ε, για τα διάφορα ταμεία και για τον προϋπολογισμό. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η πληθώρα συνεδριάσεων και βλέπουμε ότι κάποιες ενέργειες είναι ασύνδετες. Και όταν μιλάμε εδώ για το συνδυασμό ανάμεσα στον ορίζοντα 2020 και τα ταμείων ΕΣΥ και μπορεί αυτό το, να το επαναλάβουμε και σε άλλους τομείς, σε άλλες συνέργειες. Τι σημαίνει ότι όλοι εργάζονται στο δικό τους τομέα, κατανοητό αυτό, και προσπαθεί να συντονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τελικά ε, οι γενικές διευθύνσεις ε, καθοδηγούν και ο συντονισμός δεν είναι τόσο προχωρημένος ώστε να έχουμε μία κατά το μέγιστο δυνατό εναρμονισμένη προσέγγιση. Τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, να κάνει ακριβώ να βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση με τις προτινόμενες στον βασικό κανονισμό αλλαγές και να συνδέσει με δια τάξεις που ισχύουν ε, ανατομέα. Υπάρχουν ε, πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα Αν επιτύχουμε συνέπεια, ένα καλά διαρθρωμένο, ομοιόμορφο πλαίσιο που θα διέπει τη συνεργασία των ταμείων, ε, διότι τελικά ο δικαιούχος δεν ενδιαφέρεται από ποια πηγή προέρχεται η χρηματοδότηση θέλει λογιστικά να είναι ε, απλές διαδικασίες για να μπορέσει να τις διαχειριστεί. Φυσικά, είναι όντως ε, τεχνικού χαρακτήρα κάποιες αλλαγές και θα χρειαστούμε την πραγματογνωμοσύνη, τη δέουσα τεχνική πραγματογνωμοσύνη για να συζητήσουμε αυτές τις αλλαγές. Σίγουρα θα είναι ρόλος κλειδί αυτός της Επιτροπής σας. λόγω της ε, βαθιάς αναπράγματογνωμοσίας σα για το εφιστάμενο πλαίσιο και ω εκ τούτου και για τις αλλαγέ. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η συνεργασία. Να πω κάποια πράγματα για τα ΕΣΥ και για το ΕΦΣΥ. για το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το σχέδιο Juncker. Έχει θέση εκεί. Κατοχυρωμένη η πολιτική συνοχή αναφέρεται ρητά ως ένα από τα εργαλεία χρηματοδότησης για την πρόθεση της ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων εργασίας και μία από τις απαιτήσεις είναι ε, να καταστήσουμε το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα ταμεία βελτιώντα τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό ούτω ή άλλω εξυπακούεται. Μετά ε, συγκροτήθηκαν τα ταμεία ΕΣΥ ως ε, μέρος του ΕΦΣΥ, ως ε, μέσο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό και υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα στους στόχους ανάμεσα στο ΕΦΣΥ και τα ταμεία ΕΣΥ. Και έχει νόημα λοιπόν, θα πρέπει στο, στη χρήση τους να είναι συμπληρωματικά αυτά τα ε, όργανα. Ε, μπορούμε να δούμε και πιο συγκεκριμένα παραδείγματα που ε, θα είναι υποφελή και για προγράμματα ε, υποδομών, όπου μπορεί να είναι ε, χρηματοδοτήσουμε από τράπεζε ε, το, το πρόγραμμα και να χρησιμοποιηθεί η μόχλευση των ιδιωτικών ταμείων, δηλαδή ως ε, εγγύηση, ως, χρηματοδοτικό, ως επιδότηση, συγγνώμη, χρηματοδοτικό, όμω να συνδυαστούν πέρα από το ΕΣ και τα ταμεία ΕΣΥ στη χρηματοδότηση για το EAF, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το blending γίνεται ακριβώς, όχι μόνο με τα ταμεία ΕΣΥ, αλλά και με τον ορίζοντα. 2020 ε, από, μέσα από τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Έχει λοιπόν νόημα να διερευνήσουμε στους με τους οποίους μπορούμε να ε, συνδυάσουμε όλες τις χρηματοδοτικές πηγές. Το ΕΦΣΥ φυσικά θα πρέπει να είναι επωφελές όχι μόνο για τις ε, πλέον ανεπτυγμένες χώρες, τις πλουσιότερες περιοχές, αλλά και για είσαι λιγότερο αναπτυγμένες και φτωχότερες. Δύσκολα θα μοχλεύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις όταν είναι υψηλό ο κίνδυνος και ένας τρόπος για να αντισταθμίσουμε αυτό το μειονέκτημα είναι ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία ΕΣΥ για να μειώσουμε αυτό το κίνδυνο και άρα να είναι ε, τα προγράμματα ενδιαφέροντα και για τους επενδυτές. Φυσικά χρειαζόμαστε και ε, δικλείδες ασφαλείας και γι' αυτό μίλησα για τα ανώτατα όρια. Αυτά γίνονται φυσικά μόνο μετά την έγκριση κατάθεσης κατάθεση διαχειριστικής αρχής. Ο συνδυασμός ταμείων ΕΣΥ και της θα συμβεί μόνο αν το κρίνει σκόπιμο η διαχειριστική αρχή και κατά αυτόν τον τρόπο διοχετεύσει τα κονδύλια στα προγράμματα. Βάσει τη στρατηγική που ακολουθούμε γενικότερα για τα προγράμματα. Για τις νέες επενδυτικές προτεραιότητες, ε, για την ε, μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Δεν είναι ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ε, ΕΡΤΕΦ e κονδύλια ήδη, το, για το, τα, κονδύλια για το κοινωνικό ταμείο τους άλλους χρησιμοποιείται ήδη για την ενσωμάτωση. Και ο Πίτροπος ε, προμηνών έγραψε στα κράτη-μέλη και τα ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσουν ε, αυτά τα κονδύλια σε κάθε ε, περίπτωση. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση προκύπτει από τη μεταναστευτική κρίση. Χρειάζεται μια σαφέστερη βάση. Εάν ε, χρησιμοποιείτε κάποια κονδύλια θα πρέπει να δείτε αν όντω υπάρχει σωστή νομική βάση. Δηλαδή ε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε μέσα από τη σαφέστερη διατύπωση. Οι διαχειριστικές αρχές ξαναλέγουν τον τελευταίο λόγο. Θα αποφασίσουν εάν μπορούν να θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιλογές επαναδιοχετεύοντας, επανακατευθύνοντας ε, ε, κάποια κονδύλια. Ξαναλέω, είναι ε, όμως ε, βοηθάει αυτό το νέο πλαίσιο αν ε, επιλέξουν αυτήν την οδό για τις υποδομές. Δεν μιλάμε τώρα για το τσέκ επιταγών, λευκών επιταγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε. Δεν υποστηρίζουμε επενδύσεις ε, ως αυτό σκοπό πρέπει να εντάσσονται σε μια στρατηγική για μια περιοχή ε, για να δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση για να επιδεχθεί η οικονομική μεγέθυνση. Για τον τουρισμό, όντω ε, μπορεί να είναι αυτό μέρο του πακέτου για την ανάπτυξη μιας περιοχής υποστηρίζοντας πολιτιστικά μνημεία, παραδείγματος χάρη, και έχουμε δει ότι προέκυψαν στο παρελθόν κάποιε ανομαλίε με ε, σε αυτόν τον τομέα. Για τις συνέργειες και πώς θα λειτουργήσουν όντως στην πράξη αυτές, αυτό το νέο εργαλείο, το SEO. Κρατικές προμήθειες είναι αυτές που είναι. Δεν πρόκειται τώρα να αλλάξουμε για την περίοδο 2014-2020 βασικές παραμέτρους ε, των διατάξεων ε, κρατικών προμηθειών είναι εφαρμοστές και για τα ταμεία αυτά θεωρούνται ως ε, δημόσια χρηματοδότηση η διατάξη όμως δεν εφαρμόζεται για την άμεση χρηματοδότηση από τον προπολογισμό μέσα από το πρόγραμμα, μέσα από τον ορίζοντα 2020 για την περίοδο μετά το 2020 μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αυτή τώρα αποκλείται να αλλάξουν οι κανόνες. Για ορισμένα σημεία τι κάναμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ε, η σφραγίδα αριστείας, ε, Φερρυπίν, ε, είναι τώρα πλέον σαφής η ερμηνεία. Δηλαδή, ε, τι γίνεται με τις κρατικές προμήθειες, δεν υπάρχει υποστήριξη για δράσεις που αναγνωρίστηκε ότι πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν υποστήριξη ορίζοντα 2020, fast tracking δηλαδή των ε, κρατικών προμηθειών ε, και επειδή είναι σε ενωσιακό επίπεδο πλέον το χρηματοδοτικό μέσο, ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να περάσουμε από τον έλεγχο των κρατικών ε, προμηθειών. Με ε, στοχευμένο τρόπο αντιμετωπίζουμε αυτή τη δυσκολία που αναφέρατε. Τώρα, όταν ε, πρόκειται για τομείς ε, κοινωνικού ταμείου περισσότερο από ότι περιφερειακών ταμείων, θα χρειαστεί να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Όταν εγκριθούν αυτές οι διατάξει, τότε ε, θα προσφέρουμε κατευθυντήρε γραμμές στα κράτη-μέλη και όντω για τους ε, θα πρέπει να κάνουμε και αυτή την παιδαγωγική δράση και θα πρέπει και αυτοί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τους ελέγχους. Τέλος. Ε, ακούστηκε κάτι ενδιαφέρον για τον ε, συνδυασμό τη συσχέτιση ελέγχου και κινδύνου. Δηλαδή να, είμαστε, να κάνουμε πιο στοχευμένα τους ελέγχους ε, στους δικαιούχους. Μα υπάρχουν δύο επίπεδα ελέγχων από τις διαχειριστικές αρχές και οικονομικός ελέγχος που έπεται. Οι διαχειριστικές αρχές ε, που ε, κάνουν τους ελέγχους όντως θα πρέπει να προσανατολίζονται στον κίνδυνο. Δεν θα πρέπει να χαλάνε το χρόνο τους ε, ελέγχοντας δικαιούς όπου ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Ο οικονομικός όμως έλεγχος τι μας διασφαλίζει το σύστημα, όχι τις συγκεκριμένες επιχείρησεις, συγκεκριμένους δικαιούς. Αν λειτουργεί ορθά το σύστημα, αυτό ελέγχουμε με τα audits. Ε, ο φορέας οικονομικού ελέγχου με πολύ περιορισμένο ε, πεδίο δράσεων ε, ε, μέσα από στατιστικά δείγματα μπορεί να επιτύχει αυτή τη διασφάλιση. Δεν αυτό αποκλείονται αυτοί οι έλεγχοι, διότι ξαναλέω πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα από στατιστική ε, πλευρά, αλλά ξαναλέω υπάρχουν ε, πολύ περιορισμένες, είναι που πρέπει να ελεγχθούν για να είναι ε, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτέλεσματα των οικονομικών ελέγχων. Timeline χρονοδιάγραμμα. διάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισπεύσουμε εδώ. Σίγουρα είναι στόχος μας μέχρι το, τα μέσα του 17 να έχουν εγκριθεί οι νέες διατάξεις. Και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να αποσκοπούν ε, όλα τα θεσμικά όργανα για να υποφεληθούμε στο μέγιστον για τα προγράμματα που θα τρέξουν μέχρι το 2020. Ευχαριστούμε. <coughs> Σας ευχαριστούμε κύριε Μάρτιν. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. <coughs> και πριν από τη συνάντηση των συντονιστών για τη μελλοντική μας δουλειά. Σας ευχαριστούμε για το έργο που επιτελέσατε, την παρουσίαση και για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας. Τώρα θα κλείσει το δημόσιο τμήμα της συνεδρίασης. Προσκαλώ όλα τα μέλη <coughs> που δεν εκπροσωπούνται στη συνάντηση συντονιστών να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Θα συνεχίσουμε με συνεδρία συντονιστών τώρα λοιπόν.